Είναι τώρα μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, ειδικότερα στις περιπτώσεις της Σακίν Μοχάμι Ταστιάνη και της Ζάρα Μπαχράμι. Και τον λόγο έχει εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Τσόλος. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, επειδή δεν μπορεί να είναι παρούσα Κάθριν Άστον, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, μετά από διαβουλεύσεις με εκείνη θα σας παρουσιάσω τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράς, Ιράν είναι θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Τους τελευταίους μήνες η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η Κάθριν Άστον <clears throat> και οι υπηρεσίες της κατ' επανάληψη μίλησαν για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Πολλοί από εσά έκαναν το ίδιο είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να καταδικάζουμε αυτές τις απάνθρωπες πρακτικές που δυστυχώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται και ακόμα στο Ιράν. Μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύσε τον περασμένο Ιόνιο κάλεσε το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης, να σεβαστεί το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και να διακόψει οποιασδήποτε διακρίσεις κατά των εθνικών μειονοτήτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των γυναικών. Η θανατική ποινή και τα δικαιώματα των μειονοτήτων αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέτος. Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν απαιτεί από το Ιράν τίποτα περισσότερο από αυτό που απαιτεί από άλλες χώρες. Καλούμε απλώς τις αρχές του Ιράν με δημόσιες δηλώσεις και με πιστευτικές επαφές μέσω διπλωματικών εκπροσώπων να σέβονται τα δικαιώματα των πολιτών κάτι το οποίο έχουν αναλάβει να κάνουν οι Ιρανοί ε, υπογράφοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλες σχετικές πράξεις. Η συνάδελφος Κάθριν Άστον και οι ε, πρόσωποι της στη Βρυξέλλες και την Τεχεράνη ε, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην υπόθεση της, της κυρίας Ακινέ Μοχάμι Ντεφιάνη και της κυρίας Ζάχρα Μπαχραμή ε, έκαναν μια ανακοίνωση στην οποία καλούσαν τις Ιρανικές ε, αρχές να ξαναδούν το θέμα της κυρίας Ταυτιανή και άλλων ατόμων που έχουν καταδικαστεί σε ποινές σε μια χώρα όπου η θανατική ποινή δυστυχώς εξακολουθεί να ισχύει νόμιμα. Το Επίσης κινήθηκε το ζήτημα μέσω διπλωματικής οδού στις Ιρανικές αρχές. Είναι τόσο βάρβαρη και η μόνη σκέψη του λιθοβολισμού που απαιτείται να επιδείξουμε όλη τη δέουσα στεναρότητα έως ότου τεθεί τέρμα σε αυτές τις πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθεία με την Ιρανική κυβέρνηση αναφέρθηκε στο θέμα της κυρίας Ζάχρα Μπαχραμή, της οποίας η σύλληψη έγινε στη διάρκεια των διαδηλώσεων που έγιναν το Δεκέμβριο του 2000 στη Διχεράνη κατά τον εορτασμό της ημέρας της Ασούρα. Επιμένουμε ότι η κυρία Χραμή, η οποία έχει και Ιρανική και Ολλανδική υπηκότητα, δικαιούται δίκαιη σε διαφανείους και ανοιχτής δίκης. Πρέπει κατά την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κυρία Μπαχραμή να τύχει κάθε προξενικής και δικαστικής υποστήριξης θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε στενή συνεργασία με την διπλωματική εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη. Εξακολουθούμε να καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν όσο υπάρχουν αυτές οι παραβιάσεις μέσω διμερών επαφών, δημόσιων ανακοινώσεων και δηλώσεων ή στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε τους ομιλητές εν ονόματι των πολιτικών ομάδων και πρώτα η κυρία Αντζελίλη για το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίθοβολισμοί, βασανιστήρια, ε, πράξεις βάρβαρες και απάνθρωπες, οι οποίες παραβιάζουν κατά τρόπο, από τρόπο τα βασικότερα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιαστούν τέτοιες πράξεις, παρά μόνο τα λόγια τη ίδια της κυρία Ακινέ. Ε, ε, της Ακινέ μάλλον, η οποία σε μια επιστολή της ε, αναρωτιέται τι γίνεται και πώς ετοιμάζονται πριν μου πριν πετάξουν πέτρες, πώς στοχεύουν και σημαδεύουν τα χέρια και τα πόδια μου. Ε, δεν καταλαβαίνουν αυτό το φόβο φόβο του θανάτου ε, θέλω να κάνω το παν για να μείνω ζωντανή. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την κραυγή απελπισία να την ακούσει το Ευρωκοινοβούλιο. Τη Σακινέ δεν μπορούμε να την αφήσουμε μόνη τη. Θα πρέπει και εμεί να προβάλλουμε τη δική μα σημαία, τη σημαία, να υψώσουμε τη σημαία τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να παρέμβει και να σταματήσει αυτή την συνοπτική εκτέλεση. Θα πρέπει να έχουμε το κουράγιο και την τόλμη να πούμε ότι μπορούμε να θέσουμε και να διακόψουμε τι διπλωματικέ μα σχέσει σε περίπτωση ε, που πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί δεν γίνονται εκπτώσει και δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι. Ελεύθερε γυναίκε και ελεύθεροι άντρε, ελεύθεροι πολίτε όπω είμαστε, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τέτοιε πράξει. Θα πρέπει να ε, στηρίξουμε την ε, κοινή γνώμη του Ιράν που διαφωνεί με το κυβερνών καθεστώ. Θα πρέπει λοιπόν να φανούμε εκεί αδιάλακτοι και ανυποχώρητοι. Τα καθεστώτα αυτά που βασίζονται στο φόβο, στην καταστολή, στην παραβίαση των ελευθεριών και των βασικών δικαιωμάτων, εκεί θα πρέπει εμείς από αυτήν την αίθουσα της Ολομέλειας να πιώσουμε τη φωνή μας και να πούμε με τρόπο ηχηρό ότι θα προστατεύσουμε την Σακινέ. Ευχαριστώ και τώρα για τους σοσιαλιστές η κυρία Μουνίστε Ουρκίζα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η μοιχεία, η ομοφιλοφιλία, η, η, ειρηνική συμμετοχή σε δηλώσει και διαδηλώσει είναι τρία δικήματα τα οποία τιμωρούνται με φρικτές ποινέ στο Ιράν. Πάρα πολλά άτομα έχουν καταδικαστεί, κάτι που δεν θα συνέβαινε αλλού και βάση περιπτώσει όχι στην Ευρώπη. Υπάρχουν άλλωστε διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων δεν μιλάμε για αδικήματα και δεν μπορούμε να καταδικάσουμε ανθρώπους μεταξύ των οποίων και ανηλίκων για ορισμένες ε, πράξεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για αδικήματα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να απαιτήσουμε να μην ε, εκτελεστεί η Σακίνε Μοχαμάντι Αστιανή να εφαρμοστεί το δικαιοστάσιο από το Ιράν και να γίνει μια αποστολή ε, του ΟΗΕ που θα επιτηρήσει την άσκηση και την ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Πρέπει να απαγορευθούν μετακινήσεις ε, των εκπροσώπων της Ιρανικής κυβέρνησης, να μην γίνονται δεκτοί στις χώρες μας οι εκπρόσωποι της Ιρανικής κυβέρνησης. Ζητούμε από το Συμβούλιο να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ και τώρα για τους φιλελευθέρους η, η κυρία Σράκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Εδώ δεν πρέπει μόνο επειδή θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινότητα αξιών και ελευθεριών και καταδικάζουμε τη θανατική ποινή να λάβουμε δράση, αλλά και επειδή γνωρίζουμε ποια είναι τα άτομα που κρυπτούν οι αριθμοί. 388 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2009 και μόνον. Η ξεχωριστή αυτή θάνατη ατόμων ήταν ε, ισοδυναμούν με κραυγέ ελευθερία, αλλά εκπροσωπούν και ένα πλήθο άλλων που έχουν εκτελέσει στο παρελθόν. Η συζήτηση λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν είναι κάτι που οργανώθηκε στο Ιράν γιατί εφορούσε πολίτε του Ιράν που ζουν στην Ολλανδία και του συγγενεί του που είναι φυλακισμένοι εκεί. Εδώ λοιπόν ε, θα πρέπει οι Ολλανδοί διπλωμάτε να ξέρουμε ότι δεν κατάφεραν να μιλήσουν με φυλακισμένου στο Ιράν, ούτε καν με του δικηγόρου του δεν μπόρεσαν να έρθουν σε επαφή. Θα πρέπει λοιπόν ασχέτω με την κάθε ξεχωριστή υπόθεση, να δούμε ποια είναι η συνταγματική υποχρέωση, να παρέχουμε προστασία σε πολίτε μα. Αυτό ε, αφορά όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με το Ιράν. Μιλάμε εδώ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να έχουν άμεση προτεραιότητα στι ατζέντε μα. Εδώ μιλάμε για άτομα, πολίτε, γυναίκε που οι ζωέ του, αν υποθέσουμε ότι ακόμη είναι ζωντανοί, μπορεί να έχουν τερματιστεί. Η Ζαράκη δεν εκπροσωπούν μόνο μερικού από του χιλιάδε φυλακισμένου στο Ιράν. Ε, Άνδρε και γυναίκε που οι φωνέ του δεν μπορούν να ακουστούν. Η κυβέρνηση του Ιράν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η στατιστική τεχνολογία, η σκληρή γλώσσα ή οι ε, αυστηρέ ποινέ δεν μπορούν παρά να οδηγήσουν τη χώρα σε απομόνωση. Δεν θα την επιτρέψουν να προοδεύσει. Και δεν εξασφαλίζεται έτσι η ευημερία των πολιτών ούτε η αξιοπιστία τη σε διεθνέ επίπεδο. Η δικαιοσύνη και η ασφάλεια είναι διόψει του νομίσματο. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να ξέρουμε ότι ε, απαγχωνίζονται παιδιά, υπάρχουν ε, ε, βιασμοί και συνεχείς ε, ποινές και τιμωρίες. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σκεφτούμε την επιβολή κυρώσεων και την ε, πίεση του Ιράν στο πιο ευαίσθητο σημείο του, τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα για τους πρασίνους η κυρία Λόχ Μπίλερ για τρία λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στα πλαίσια της ε, καταδίκης των ε, δύο γυναικών έχουν ε, ήδη εξηγηθεί οι λόγοι και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ιράν μία κίνηση ε, για, ε, κατά αυτών των τρομερών ε, πράξεων και υπάρχει μία κίνηση ο Αγιατόλα Σαράουντι πρώην επικεφαλής στα θέματα δικαιοσύνης είχε καταδικάσει ήδη το 2008 και ε, δίνει το, τη δυνατότητα η τοπική νομοθεσία να ε, πάρει μία απόφαση ένας δικαστής και ε, είχε αρθεί πέρυσι τον Ιούνιο το άρθρο σχετικά με τους λιθοβολισμούς μέχρι ότου το θέμα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο. Άρα πρέπει αυτά να γίνονται σεβαστά. Βέβαια το Νότα το δικαστήριο εξετάζει εάν συνάδουν με τον νόμο αυτές οι πράξεις και ε, απαγορεύονται οι λιθοβολισμοί. Θα μπορούσε όμως το δικαστήριο αυτό να επαναφέρει τους λιθοβολισμούς. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν ε, για να απαγορεύσει τους λιθοβολισμούς και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία έκκληση εις ε, το Κοινοβούλιο διότι ο στόχος μας είναι να σωθεί η σακινέ Μοχαμάτι Αστιάνη. Μπορεί στο τέλος να μην λιθοβοληθεί αλλά θα μπορούσε ε, να καταδικαστεί ε, το να την ε, κρεμάσουν. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει μία πιο εκτενής νομική εξέταση της περιπτώσεώς της. Είναι κάτι που θα έπρεπε να αρχίσει ήδη και πολύ σωστά η κυρία Άστον ζήτησε ζήτησε να αναλυφθεί αυτή η δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος και τώρα για τους Ευρωπαίους ε, ε, Ευρωπαίους μιλάει ο κύριος Τάνοκ. Ακόμα μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ε, με το Ιράν που εκτελεί, εκτελεί παιδιά, λιθοβολεί γυναίκες επειδή ήταν Μιχαλίδες και επιβάλλει τη θανατική ποινή οι άλλες χώρες, ε, οι λίγες που υπάρχουν ακόμα που εφαρμόζουν θανατική ποινή, ε, την εφαρμόζουν μόνο για δεχθεί εγκλήματα. Κάτι που δεν ισχύει καθόλου στο Ιράν. Ένα αγόρι 16 ετών δεν είχε επιτεθεί σε κανέναν ούτε εν τον ομοφιλόφιλος. Παρόλα τα αυτά ο δικηγόρος του ο Μουστάφη χρειάστηκε να αρχίζει να κρύβεται διότι κινδύνευε να συλληφθεί. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση της Ξακινέ Αστιάνη η οποία κατηγορείται για μοιχεία διαφθορά επειδή κυκλοφόρησε, εμφανίστηκε χωρίς κάλυμα της κεφαλής σε ένα ξένο περιοδικό και τώρα ε, κατηγορείται ότι ήταν συνένοχος σε ένα έγκλημα το οποίο υποχρεώθηκε, υποχρεώθηκε να παραδεχθεί. Πρέπει λοιπόν να καταδικάζουμε τις παραβιάς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν σε κάθε περίπτωση όπως καταγγέλουμε το πυρηνικό του πρόγραμμα και μην ξεχνάμε και την περίπτωση της σύλληψης της κυρίας Μπαχράμι που έχει διπλή Ιρανική και Ολλανδική υπηκότητα. Καλούμε λοιπόν μέσω του Κοινοβουλίου στον πρόεδρο του Ιράν να επιδείξει επίοικια χωρίς δυστυχώς πολλές ελπίδες. Ευχαριστώ και τώρα για την ε, ε, ομάδα της, Επιτρο... της Ηνωμένης Αριστεράς ο κύριος Ζάκη Ενάν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι διαμαρτυρίε και τι ανησυχίε που εκφράζονται για την ε, ελευθερία στο Ιράν. Θα ε, στηρίξουμε όλου του δημοκράτε που θέλουν η δικαιοσύνη να αποκτήσει νόημα. Εδώ λοιπόν χειρά καταδικάζουμε την ε, καταδίκη και την σύλληψη την ίδια τη κυρία Αστιάνη. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ούτε την επιβολή τη ποινή ούτε τον λιθοφολισμό. Θέλουμε την απελευθέρωσή τη. Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα κράτη που έχουν τον λαϊκό κοσμικό χαρακτήρα ως αρχή τους και τον κοσμικό μάλλον χαρακτήρα ως αρχή του και πρώτη του αξία να εμποδίσουν αυτήν την ε, δολοφονία της ίδια της ελευθερίας, τη ε, της δημοκρατίας να καταργηθεί η θανατική ποινή σε όλες τις χώρες. Εδώ θα πρέπει λοιπόν οι δικαστικές αρχές του Ιράν να επιβάλλουν ε, μορατόριο για την υλοποίηση της θανατικής ποινής. Να μην χρησιμοποιούνται τέτοιε ποινέ όπω λιθοβολισμοί και τα βασανιστήρια σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο. Ευχαριστώ και τώρα για την Ευρώπη τη Ελευθερία και τη δημοκρατία ο κύριο Περών για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με όλους όσοι είπαν ότι δεν θα πρέπει να εξακολουθήσουν αυτές οι βαρβαρότητες όπως ο λιθοβολισμός για μοιχεία. Θα πρέπει εδώ να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα και της Ακινέ και όλων των γυναικών και των ανδρών που βρίσκονται στην ίδια θέση. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστό, σεβαστά τα ανθρώπινά τους δικαιώματα. Θα πρέπει εδώ να προγραμμίσω κάτι που το άκουσα μία φορά μόνον, αλλά από τον τελευταίο συγκεκριμένα αγορητή. Ε, πολλά από αυτά που σήμερα ε, αντιμετωπίζουμε προκύπτουν από την ε, γενιά των θρησκευτικών εξτρεμιστών οι οποίοι είναι φονταμενταλιστές ως προς την εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου. Εδώ λοιπόν φαίνεται να υπάρχουν τέτοιε τάσει παρίσφυσης και στη δική μας ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη. Ευχαριστώ και τώρα ερχόμαστε στου επόμενου ε, εγγεγραμμένου ομιλητέ, η κυρία Μαντσόνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που ε, με την ε, σχεδόν ομόφωνη ψηφοφορία ενέκρινε την διοργάνωση της συζήτησης αυτή για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Η δική μου η έκκληση που υποβάλλω μαζί με την συνάδελφο Αλτζελίλη προσυπογράφηκε από πολλού συναδέλφου του Ευρωκοινοβουλίου με την ελπίδα να, να σώσουμε μία ζωή. Διότι η σημερινή μέρα για τη Σακινέ μπορεί να είναι η τελευταία και ίσω ε, και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο ε, γιατί η δική μας η έκκληση ξεπερνάει κάποια όρια. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η περίπτωση αυτής της γυναίκας εκφράζει τις περιπτώσεις πολλών άλλων γυναικών, ανδρών και νεαρών ε, πολιτών στο Ιράν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Το καθεστώς καταπατά τις ελευθερίες των γυναικών και κυρίως αγνοεί τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν έχει εγκρίνει ψηφίσματα για δύο τέτοιες υποθέσεις τον περασμένο χρόνο και για τις σχέσεις με, την, με το Ιράν και ήδη υπήρξαν δύο τοποθετήσεις τον ε, Ιούνιο και τον Ιούλιο φέτος και ο ΙΕ ενέκρινε ψηφίσματα ζητώντας την ε, άρση της θανατικής ποινής, την κατάργησή της, την πλήρη θεωρώντας ότι το η Ιράν θα πρέπει να συμμετάσχει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητηθούν τα δικαιώματα των γυναικών. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ του ίδιου για την προστασία των γυναικών. Όμω η κυβέρνηση του Ιράν φαίνεται να λέει ότι αν θέλετε να συζητήσετε μαζί μα, εμεί αυτοί είμαστε και αν σα αρέσουμε. Ε, Όμω η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πυλώνα τη εξωτερική πολιτική τη Ένωση. Και αυτό μα καλεί να αναλάβουμε τι ευθύνε μα ω γεγονό. Θα πρέπει λοιπόν να τι αναλάβουμε και σε σχέση με παρόμοιε υποθέσει που μπορούν να θέσουν εν κινδύνο και την διαδικασία ενσωμάτωση. Όλε οι εθνικέ κυβερνήσει έχουν κινητοποιηθεί και θα πρέπει και εμεί από πλευρά μα να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Οι νέοι Ιρανοί σε διαδήλωση που οργανώθηκε στην Ιταλία είπαν ότι δεν πιστεύουμε ότι, μπορού, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Μπορεί να σώσουμε μια ζωή, αλλά δεν θα σώσουμε το Ιράν. Εμεί με σοβαρέ κυρώσει και ποινέ θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτή η κινητοποίηση είναι μόνο το πρώτο βήμα και ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την οδό και θα φτάσουμε μέχρι και σε εμπάργκο, μέχρι και σε διακοπή των σχέσεών μα με το Ιράν, αν χρειαστεί. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Κώστα για 1,5 λεπτό λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με αυτή τη συζήτηση που ειλικρινώ ε, πίστευα ότι θα είχε μεγαλύτερη συμμετοχή, γιατί τη αξίζει αυτή η συμμετοχή, ε, θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή μου σε όσε ακούστηκαν και σε όσου κινητοποιήθηκαν τι τελευταίε ημέρε σε διεθνέ επίπεδο. Διότι η καταδίκη σε θάνατο τη Σακινέα Τάνη ε, και βεβαίω μετά από την έκκληση του γιού τη του Σαΐντ για να σωθεί και η ίδια αλλά και τόσε άλλε γυναίκε που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο, όπω η κυρία Ζαρά Εμπαράνη και τόσε άλλε που έχουν καταδικαστεί, είναι υποθέσει που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, πολιτών είναι δύο θέματα αδιαίρετα, ε, Πρέπει να τα δούμε από κοινού. Πρέπει να προστατεύσουμε και τι δικέ μα συνειδήσει και ελευθερία, την ελευθερία μα, σώζοντα τι γυναίκε αυτέ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, ε, θα πρέπει και ο Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η κυρία Ρέντινγκ, να κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα, όπω ήδη έχουν κάνει, ενώπιον τη Ιρανική κυβέρνηση και σε διεθνέ επίπεδο, ώστε η δική μα κινητοποίηση για την απελευθέρωση τη Ακρά, για την μη επιβολή τη ποινή τη Ακινέ, για την κατάργηση των λιθοβολισμών να εξακολουθήσουν, να κινητοποιηθούμε για να καταργηθεί η θανατική πηδή και να στηρίξουμε τη δημοκρατισμό του Ιράν. Στο, σε ιταλικό επίπεδο, όλοι οι συνάδελφοι έχουμε οργανώσει εδώ, στο χώρο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ε, στο Στρασβούργο μία ε, ε, εκδήλωση που ονομάζεται Φω για τη ζωή τη Σακινέ. Καλούμε όλου του συναδέλφου να συμμετάσχουν γιατί αυτή η τραγική υπόθεση που είναι τόσο χαρακτηριστική δεν θα τελειώσει εδώ. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε μόνο το ταφό των ε, λαό ούτε του αντιφρονούντε του Ιράν. Θα πρέπει να έχουμε ισχυρότερη παρέμβαση από την πλευρά τη Ένωση διότι θεωρούμε ότι για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ στον κόσμο μα ε, ε, κρίνονται η αξιοπιστία και το κύριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Κιλ Νίσερ για τους πράσινους. Η περίπτωση της Σακινέ η οποία μας έχει κινητοποιήσει και εμάς και πολλούς πολίτες στην Ευρώπη μας ε, αναγκάζουν να θυμηθούμε την περίπτωση και άλλων γυναικών και σκέφτομαι τη Ζάρα Μπαράμι η οποία βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση απειλείται με εκτέλεση μετά από μια δίγη που έγινε κάτω από παρόμοιες συνθήκες πιέσεις δηλαδή απομόνωση για πολλούς μήνες απόλυτη απομόνωση βασανιστήρια για να ομολογήσει πράγματα που κατόπιν δεν αναγνωρίζονται χωρίς ε, την παρουσία δικηγόρων, χωρίς ε, υπεράσπιση. Υπάρχει και η περίπτωση του Μπρέιμ Αμιντή που αναφέρθηκε προηγουμένως, ενός ανηλίκου που και εκείνο δεν έχει δικηγόρο, ή της Σιβάνα Ζαράρη, δημοσιογράφου που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Amnesty International τη θεωρεί σαν ε, φυλακισμένη για λόγους πεπιθήσεων, η οποία είναι κλεισμένη, φυλακισμένη σε ένα κλουβί όπου δεν μπορεί να κουνήσει ούτε τα πόδια τα χέρια και αυτή απειλείται με εκτέλεση. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε για τη Σακινέα και για όλες ε, τις περιπτώσεις αυτές να απαιτήσουμε την ε, δικαιοστάσιο, μορατόριου για όλες τις εκτελέσεις, την κατάρριξη της θανατικής ποινής, ε, και να μην ε, πάθουν τίποτε όσοι συμμετέχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις, να προστατεύονται οι ανήλικοι και απαιτούμε οι εκπρόσωποι του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού να μπορέσουν να επισκεφθούν τις κρατούμενες στη φυλακή. Ο κύριος Ρώση τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τις τελευταίες ημέρες πολλοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικοί διανοούμενοι, και εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας ε, κινητοποιήθηκαν για την απελευθέρωση της Ακινέ. Ε, μια Ιρανή μητέρα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο ε, διαλυθοβολισμού επειδή διέπραξε μοιχεία και επειδή της αποσπάσαν ε, μια ε, παραδοχή της ενοχής της ε, είναι κάτι το απαράδεκτο. Αυτό είναι μια μορφή βασανιστηρίου. Το θύμα αυτό πρέπει να λιθοβοληστεί μέχρι να πέσει νεκρό στο έδαφος με το κεφάλι. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι δεν, μπορούμε να, δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος τέτοιου θανάτος και λιθοβολισμού που να, ε, ακαριέως να επιφέρει το θάνατο. Γίνεται σταδιακά αυτό και μπορεί να θεωρηθεί μορφή βασανιστηρίου. Και αυτό έχει συμβεί με πολλές γυναίκες στο Ιράν που θεωρείται ότι έχουν διαπράξει Τουλάχιστον 40 γυναίκε είναι φυλακισμένε, περιμένοντα και αυτέ να θανατωθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι λοιπόν αναγκαία η, παρέμβαση του Κοινοβουλίου να υψώσουμε τη φωνή μα για να σταματήσουν αυτέ οι βαρβαρότητε. Ευχαριστώ τώρα η κυρία Στρίφλερ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, σας εκπροσωπώ εδώ τη Ρασίντα Ντατή, η οποία συνέταξε το ψήφασμα, ψήφισμα εν ονόματι του ΕΛΚ και δυστυχώς είναι στο Παρίσι σήμερα. Έγινε το ψήφισμα αυτό για δύο λόγους. Αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να υψώψει τη φωνή του μαζί με τις διεθνείς οργανώσεις, τις κυβερνήσεις και όσους υπερασπίζονται τη Σακινή και το ε, την ε, Σακινέ Μωαμάρα Στανή και αντιτίθεται τίθενται στην θανάτωσή της διαλυθοβολισμού. Μία ε, γυναίκα η οποία ήταν πάντοτε προπομπός στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορεί να σιωπήσει και να αφήσει να σκοτώσουν την ε, Σακινέ. Δεν είναι παρέμβαση να επιθυμίζουμε σε όλους ε, ότι έχουμε μία κοινή κληρονομιά και αξίες και δεύτερον η διάζουσα σε περίπτωση της Σαγκινέ οδήγησε τη Ρασίδα Ντατή να θελήσει να υψώσει τη φωνή της κατά όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και θυμάτων της βίας και στη συνέχεια αναφέρουμε και την Τζάρα Μπαραμή της Ολλανδέζας η οποία συνελήφθη στο Ιράν και υποχρεώθηκε ε, να ομολογήσει τις κατηγορίες εναντίον της και να τις αποδεχθεί στην τηλεόραση. Πρόκειται για γυναίκες που δεν μπορούν πλέον να αμυνθούν και να ονόματι της κυρίας Ρασίντα Ντατή παρακαλώ να υπερψηφίσετε για να αντιταχθείτε σε μια τέτοια ε, καταδίκη. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γκόμες για 1,5 λεπτό. Τα άτομα αυτά είναι ακόμη μερικά από τα χιλιάδες θύματα του Ιρανικού καθεστώτος. Η κυρία Μπαχράμι, η Σακινέ, είναι γυναίκες που κινδυνεύουν από λιθοβολισμό. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα αυτή δεν είναι μέλο του Συμφώνου για την Σταθερότητα και την Προστασία των Ανθρωπίνων Ελευθεριών. Αυτά λοιπόν είναι πράξει που αμαυρώνουν την φήμη του μεγάλου Ιρανικού πολιτισμού στη Λισαβόνα. Διοργανώθηκε ε, διαδήλω, κινητοποίηση ε, με συμμετοχή πολλών ατόμων για την ε, ε, απελευθέρωση της Σακινέ με συμμετόχους ε, και εκπροσώπους και της Βραζιλίας με, και εδώ υψώθηκαν φωνές ανθρωπιάς ε, και αλληλεγγύης υπέρ της Σακινέ. Το Ιράν το μεγαλύτερο, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο Κοινοβούλιο αύριο με τον εξή τρόπο, Πρόεδρε. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες δράσεις ώστε οι Ιρανοί να μην μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν οι ανθρώπινε ελευθερίε δεν γίνονται σεβαστέ στη χώρα του. Θα πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύουν αποτελεσματικά όσου μάχονται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Αυτό έχει σχέση με την πραγματικότητα του Ιράν. Διότι εμεί στην Ευρώπη δεν μπορούμε να μην προασπιζόμαστε αξίε οι οποίε δεν είναι πλέον μόνο ευρωπαϊκέ, είναι οικουμενικέ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι βασικέ ελευθερίε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Καρβάλιο για ένα λεπτό. Κυρία, κυρία Πρόεδρε, η Σακινέ και ε, οι παρόμοιε περιπτώσει αυτών των γυναικών αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των βασικών κοινωνικών ελευθεριών. Θα πρέπει να ενώσουμε εδώ τι φωνέ μα με όλα τα εθνικά κινήματα στήριξη των γυναικών αυτών που ζητούν την άμεση απελευθέρωση τη Σακινέ. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε ότι η ισότητα των δικαιωμάτων των γυναικών, η ελευθερία τη έκφραση και η ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών δεν γίνονται σεβαστοί στη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να προστατεύσουμε τις γυναίκες του Ιράν, να τις στηρίξουμε, γιατί ο ρόλος του στον εκδημοκρατισμό του Ιράν είναι σημαντικός. Θα πρέπει το θάρρος και το τόλμη τους να είναι στοιχεία που θα τα χαιρετήσουμε, διότι μας εμπνέουν και ο αγώνας αυτός για τη δημοκρατία και το μέλλον του Ιράν ως μιας ειρηνικής χώρας με, δικαιω... με ισότητα των δικαιωμάτων είναι αυτά που οι γυναίκες αυτές μάχονται να καταφέρουν. Ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία Catch the Eye και ως συνήθως έχουμε πολύ περισσότερους συναδέλφους που θέλουν το λόγο από ότι έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και για να μπορέσουμε να σεβαστούμε τη μερίσια διάταξη. Θα πάρω μόνο πέντε και η πρώτη είναι η κυρία Κολάνσκα Μποβίνσκα. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να καταδικάσουμε όλοι αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Είναι σημαντικό αυτό, διότι έτσι θα σώσουμε ζωές ανθρώπων. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην αντιπολίτευση στο Ιράν που θα αποκτήσει περισσότερο θάρρος για να συνεχίσει τον αγώνα της πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη δράση που αναλαμβάνουμε. Ψηφι... Θεσπίζουμε ψηφίσματα, έχουμε συζητήσει Η κυρία Άστον ε, λαμβάνει, ε, ε, κάνει διάφορες ενέργειες, διάφορα διαβήματα, χωρί όμω οποιαδήποτε απάντηση στι κινήσει που κάνουμε εμεί. Αν θέλουμε να θεωρηθούμε σαν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αγωνίζεται και προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο, αν θέλουμε θέλουμε αυτά που λέμε και κάνουμε να είναι αποτελεσματικά, πρέπει να αφιερώσουμε μια ειδική συζήτηση σε αυτό το θέμα. Να σκεφτούμε συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαμε να αναλάβουμε ώστε να έχουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριο Σταραμπέλα για ένα λεπτό προτείνω να λιθοβολήσουμε το Ιράν διότι πώς μπορούμε να δεχθούμε μια τέτοια βάρβερη ε, αντιμετώπιση του ατόμου διότι όταν ε, ε, λιθοβολείται ένας άνδρας καλύπτεται μέχρι τη μέση ενώ η γυναίκα μέχρι το στήθος από εδώ φαίνεται και δεν πρέπει η πέτρα να είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή μικρή, να μην ε, πρόκειται για βότσαλο δηλαδή. Και ε, ε, διαρκεί αυτή η διαδικασία μισή ώρα. Λέγεται ότι δεν μπορεί κανείς να υβρίσει τον υπεύθυνο και δεν μπορεί ούτε να καταφερθεί εναντίον του μετά το θάνατό του. Τι μπορούμε να κάνουμε για την κυρία Αμαντή. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει ζητήσει να της δοθεί άσυλο στην Ευρώπη και θα έπρεπε να προσθεθεί. Ο κύριος Μπιλμπάου Μπαρανίσα τώρα. Η κυρία, με συγχωρείτε. <clears throat> Πρέπει να καταδικάσουμε αποφασιστικά το Ιράν. Το Ραμαντάνι τελειώνει. πρέπει να υιοθετήσουμε μία πολύ στεναρή και αυστηρή στάση ώστε να μην εκτελέσει το Ιράν τη θανατική ποινή. Πρέπει κάθε ευρωβουλευτής και κάθε ευρωβουλευτή να μεμονωμένα να κάνουν κάθε προσπάθεια για να θέσουμε επιτέλους τέρμα σε τέτοιες βαρβαρότητες. Και καλώ την κυρία Άστον να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σεβασμό από το Ιράν των διεθνών συμβάσεων. Πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικά μέτρα και πιέσεις στο Ιράν ώστε επιτέλους να σεβαστεί τις διεθνείς συμβάσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, ασχολούμαι με τα δικαιώματα του ανθρώπου και ε, της γυναίκας γιατί είμαι νομικός, ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και 20 ε, χρόνια ε, και έχω γράψει δύο βιβλία για το θέμα αυτό και καταδικάζω κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων οποιασδήποτε γυναίκας αλλά θα έλεγα να μην πάει κάποιος στο Ιράν αλλά να έρθει στην Ουγγαρία η κυρία Άστον και να μας πει ε, ποιες είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία. Από όταν εγώ ήρθα τουλάχιστον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνω ότι μιλάμε για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουγγαρία υπάρχουν παρεμφερείς ενέργειες ε, η αστυνομία με συγχωρείτε, ε, έχει λήξει ο χρόνος ομιλίας σας και πρέπει να σας διακόψω, λέει η Πρόεδρος. Και τελευταίος, η, τελευταία η κυρία Ματέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, το να περασπιστούμε τη Σακινέ σημαίνει ότι θα περασπιστούμε τη ζωή, το δικαίωμα στη ζωή. Άρα το να μένει κανεί ζωντανό η Χάρτα των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όλε τι ταγματικέ χάρτε των χωρών μα ουσιαστικά διατρανώνουν τι αρχέ αυτέ και τα παραβία στα δικαιώματα του ατόμου. Ε, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στη ζωή κατά πρώτο λόγο. Η μάχη μα λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι μάχη για ένα μόνο άτομο αλλά για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα στου οποίου στερούν τη ζωή του σε κάθε μέρο του πλανήτη και για οποιοδήποτε λόγο. Για κανένα κανένα λοιπόν λόγο, με καμία θρησκεία ή ιδεολογία ή αρχή ως πρόσχημα, δεν μπορούμε να δεχόμαστε την καταπάτηση της ζωής ενός ατόμου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρχουν ε, δράσεις αποφασιστικές και αντιμετωπίση στεναρή των χωρών που επιβάλλουν την ε, θανατική ποινή και παραβιάζουν τις ανθρώπινες και ατομικές ελευθερίες. Εδώ θα πρέπει να είναι αποφασιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να διακόψει αν χρειάζεται τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με τέτοιες χώρες προκειμένου να γίνονται σεβαστά αυτά τα δικαιώματα. Η Σακινέ ναι, ε, δεν θα είναι μόνο το πρώτο βήμα και τώρα θα πρέπει να πούμε φτάνει αρκετά. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση έχει και άλλη το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος κύριος Τσόλος. Κυρία Πρόεδρε, Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για αυτή τη συζήτηση, για την υποστήριξη που επιδείξατε όλοι σαφέστατα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εξ ονόματος της Επιτροπής σας διαβεβαιώ ότι κάθε τι το δυνατό θα γίνει ώστε οι Ιρανικές αρχές να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο διπλωματικών συζητήσεων και η κυρία Άστον σας διαβεβαιώ δεν θα περιοριστεί σε δημόσιες δηλώσεις σας ενημερώνω ότι μία τελευταία συνάντηση ανάμεσα στην τοπική εκπροσώπηση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιρανικής κυβέρνησης έγινε στις 29 Αυγούστου η Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος θα συνεχίσει τα διαβήματα ώστε να μην εκτελεστεί η θανατική ποινή. Ευχαριστώ πολύ. Έληξε η συζήτηση. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι τώρα οι δηλώσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 105 του κανονισμού και οι ομιλητές βεβαίως πρέπει να γνωρίζουν πως ε, ως συνήθως είναι περιορισμένος ο χρόνος γιατί έχουμε πολλούς ενδιαφερόμενους. Πρώτα απ' όλα τον λόγο λοιπόν έχει η κυρία